Οι αρμόδιες ουγγρικές αρχές <clears throat> μου έστειλαν μια αίτηση για την άση της ε, ασυλίας του κυρίου Τσάμπα Μολνάρ μέσα στα πλαίσια μιας ποινική διαδικασίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η αίτηση αυτά παραπεμφθεί στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Στις 15